Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Εθνικές στρατηγικές για την αποδοτικότητα των εναλλακτικών στρατηγικών στον τομέα της ενέργειας να υπενθύσω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία έκανε πρόσφατα η Επίτροπή μας για την προμήθεια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει κατελάχιστον το ποσοστό των 35% των ανανεώσιμων πηγών και της κατανάλωσης ενέργειας και ασφαλούς κατανάλωσης ενέργειας ως δικαιώματος. Η Επιτροπή μας ε, πήρε και αποφάσεις σε σχέση με την αποδοτικότητα στον τομέα της ενέργειας. Υπήρξαν δεσμευτικοί στόχοι 35% βελτίωσης. Δεν αναφέρομαι εδώ σε εθνικούς στόχους και η, επιτροπή που ψηφί... η έκθεση την οποία ψηφίσαμε χθε στον τομέα της οικοδομής έχει σαν στόχο μακροπρόθεσμα την απανθρακοποίηση του μίξ ενέργειας που καταναλώνεται. Λοιπόν, η αποδοτικότητα της ενέργειας στα κτίρια, στρατηγικές ανακαίνησης, συνεισφορά του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, και ε, ασφαλής παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σε μισή ώρα θα έρθει ο τακτικός ε, πρόεδρος μας. Οι παρουσιάσεις ε, θα γίνουν από πέντε εμπειρογνώμονες και μετά από την παρουσίαση από τους εμπειρογνώμονες αυτούς θα υπάρξουν ερωταπαντήσεις. Οι παρουσιάσεις θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ήτρε με περιλήψεις. Ελπίζω να είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι παρακολουθούν αυτά τα οποία θα υποθούν εδώ και να μην είναι μόνο οι παρόντες. Οκτώ λεπτά ομιλία ο κάθε ομιλητής. Να θυμίσω και τους εμπειρογνώμονες ε, ότι πρέπει να σεβαστούν τον χρόνο που έχουν στην διάθεσή τους για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το πρόγραμμά μας σωστά. Πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Ντόλφ Γκίλεν που θα αναφερθεί στις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη-μέλη με στόχο την επίτευξη των στόχων για την αποδοτικότητα της ενέργειας που χρησιμοποιείται. Ο κύριος Γκίλεν είναι διευθυντής της ΑΙΡΙΝΑ από το 2011. Είναι υπεύθυνος για τις εργασίες της υπηρεσίας αυτής, λειτουργεί ως σύμβουλος η υπηρεσία αυτή σε κράτη, περιφέρειες, ε, ενέργεια, προγραμματισμό στον τομέα της ενέργειας και τα λοιπά. Πριν πάει στο Αϊρίνα, ο Γκίλεν ήταν υπεύθυνο στην οργάνωση βιομηχανικής παραγωγής των Ηνωμένων Εθνών. Κύριε Γκίλεν, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, με χαρά βρίσκομαι ανάμεσά σας σήμερα θα ήθελα <clears throat> ξεκινώντας να θέσω το πλαίσιο της συζήτησης που θα ακολουθήσουν και οι επόμενοι ομιλητές. Βασικά θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχουν ε, συνέργειες ανάμεσα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αποδοτικότητα της ενέργειας, όχι μόνο στην οικοδομή αλλά και στις μεταφορές. Ε, οι ανανεώσιμες πηγές μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε όλους τους τομείς έτσι ώστε ε, η ίδια ποσότητα ανανεώσιμων να καλύψει μεγαλύτερο τμήμα των αναγκών. Αυτό το οποίο έχουμε σαν στόχο είναι να μειώσουμε τις εκπομπές καυσαερίων και αυτό ε, ταυτόχρονα να γίνεται και σε σημαντικό ποσοστό αλλά και με σημαντικά χαμηλό κόστος. Υπάρχουν πολλαπλές ε, ε, πιθανές εναλλακτικές πηγές όπως η αιωλική, η ηλιακή κτλ. και όλες μπορούν να βοηθήσουν να πετύχουμε τις συνέργειες αυτές. Ξεκινήσαμε μία μελέτη τη Δευτέρα εδώ στις Βρυξέλλες και είδαμε ότι υπάρχει τουλάχιστον δυνατότητα κατά 34% βελτίωσης της αποδοτικότητας της χρήσης των πηγών των εναλλακτικών ενέργειας. Σχετικά τώρα με τη βελτίωση των πολιτικών θα πρέπει να έχουν σαν στόχο τις υποδομές όπως σαν παράδειγμα υποδομές για την πλήρωση των συσσωρευτών των ηλεκτροκίνητων οχημάτων στον τομέα των κατοικιών, της οικοδομής μάλλον, θα πρέπει να δούμε επίσης αν υπάρχει δυνατότητα χρήσης ε, νέων συστημάτων ανακαίνησης, εξυγχρονισμού, ε, σαν παράδειγμα θερμοπομπών, όπως επίσης ε, και όλα αυτά να γίνονται με μικρή οικονομική επιβάρυνση και όλα αυτά δείχνουν την ύπαρξη πολιτικών που έχουν σαν στόχο τη βελτιστοποίηση των χρησιμοποιούμενων συστημάτων. Θεωρούμε ότι το 90% της μείωσης των καυσαερίων που απαιτείται να πετύχουμε μέχρι το 2050 μπορεί να γίνει μέσω της αύξησης αποδοτικότητας της εναλλακτικής παραγωγής ενέργειας. Βλέπετε το μπλε χρώμα στον πίνακα. Το ποσοστό των ανανεώσιμων θα πρέπει να αυξηθεί και να φτάσει το 65% των πρωτογενών προμηθειών ενέργειας. Αυτό είναι το πράσινο κομμάτι του ε, πίνακα. Σήμερα είναι το 15% περίπου. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται αύξηση κατά 1,4 χρήση εναλλακτικών κατέτων, ενώ τώρα είναι 0,2 κατέτων. Απαιτείται ένας επταπλασιασμός ουσιαστικά της συνολικής προσπάθειας για την αύξηση των ανανεώσιμων. Θέλουμε λοιπόν 2,5 με 2,6% ετήσια τουλάχιστον βελτίωση. Στον τομέα της αποδοτικότητας λοιπόν έχουμε ένα μεγάλο κενό να καλύψουμε. Όπως είπα χτες την Δευτέρα ξεκινήσαμε ε, την έρευνα για τις προοπτικές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ε, καταλήγουμε στο ότι μπορούμε να φτάσουμε σε υψηλότερα επίπεδα και είμαστε πάρα πολύ κοντά στις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω του συμπεράσματος των 34% που έχουμε προβλέψει. Αν δείτε τα κενά τα οποία πρέπει να καλυφθούν, είναι η λεγόμενη φαιά περιοχή στον πίνακα. Βλέπετε τρεις κατηγορίες επιλογών, καταρχάς ισχυρές εξοικονομήσεις πιστώσεων, ε, μετριοπαθείς εξοικονομήσεις και επιπλέον κόστος. Ε, συνδυασμός αποδοτικότητας και ανανεώσιμων, ηλεκτροκίνηση, θερμοπομπή, όλα αυτά είναι στις λεγόμενες ενδιάμεσες κατηγορίες. Εξετάσαμε λοιπόν τις δυνατότητες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με ε, στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας κατά 30%. Υπάρχουν και άλλες μελέτες εκτός της δικής μας που λέγουν ότι υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης που φτάνουν και το 35%. Πάντως με το 30% πετυχαίνουμε το 34% στα ανανεώσιμα, με 35% βελτίωση αποδοτικότητας φτάνουμε σε 37% χρήσης εναλλακτικών. Βλέπετε λοιπόν την ανάγκη για συνέργειες ανάμεσα στους δύο κλάδους. Έχουμε κάνει λεπτομερείς επίσης αναλύσεις ε, για τις ε, διάφορες οικονομικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται. Βλέπουμε στην Γερμανία σαν παράδειγμα, αναχώρα, βλέπουμε ότι υπάρχουν θετικές συνέργειες αντίστοιχες καταρχάς από χώρα σε χώρα παρά τις κάποιες διαφορές. Όσο υψηλότερη είναι η αποδοτικότητα, τόσο υψηλότερο είναι πάντα και το ποσοστό των ανανεώσιμων το οποίο μπορεί να ανοιχνευτεί. Η αποδοτικότητα βοηθάει λοιπόν τις ανανεώσιμες, αλλά και οι ανανεώσιμες βοηθούν την βελτίωση της αποδοτικότητας. Αυτό φαίνεται σε αυτόν τον πίνακα. Συνολικά μπορούμε να πούμε ότι περίπου το 1 τέταρτο της, αποδο, βελτίωσης αποδοτικότητας εξαρτάται από την επιταχυμένη θα έλεγα εφαρμογή των ανανεώσιμων, ιδιαίτερα τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας για τον τομέα των μεταφορών. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Οι δυνατότητες λοιπόν από τη μία βρίσκονται στην χρήση περαιτέρω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πολλές από τις επιλογές υπολογίζονται με στόχο το 100%. Αν το συνδυάσει κανείς αυτό με την υψηλή αποδοτικότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται και με την δυνατότητα χρήσης στην αυτοκίνηση, βλέπουμε ότι μπορεί να έχουμε πάρα πολλά κέρδη στον τομέα αυτό. Το ίδιο ισχύει και κυρίως και στην υδροηλεκτρική και στην αιωλική και στην ε, ηλεκτρική παραγωγή και ε, επίσης με διαφορετικά επίπεδα στη γεωθερμία ε, και σε άλλους τρόπους παραγωγής ενέργειας όπως η βιομάζα κτλ. Λοιπόν, αυτά είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω τεχνικές λεπτομέρειες. Ευχαριστώ κύριε Ντίλον, ευχαριστώ που σεβαστήκατε και τον χρόνο που είχατε στη διάθεσή σας. Με χαρά τώρα θα ήθελα να σας παρουσιάσω τον την κυρία Κριστιάνη Έγκερ. Θα σας μιλήσει για το benchmarking στα κράτη-μέλη και τις εθνικές στρατηγικές αποδοτικότητας της ενέργειας. Η κυρία Έγκερ είναι υπεύθυνη για θέματα ενέργειας της ΟΕ, Αυστριακής Υπηρεσίας Ενέργειας της Βόρειας Αυστρίας. Και είναι μάνατζερ επίσης ε, ενός επιχειρηματικού δικτύου 142 επιχειρήσεων που απασχολούνται στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας και των ανανεώσιμων πηγών. Είναι αντιπρόεδρος και του Φιντερίν του Ευρωπαϊκού Δικτύου Περιφερειακής Ενέργειας και περιβάλλοντος. Είναι επίσης και η Conference Director ε, μιας από τις πιο σημαντικές συναντήσεις σε αιτήσια βάση για την αποδοτικότητα της ενέργειας στην Ευρώπη. Κυρία Έγκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους. Αυτά τα οποία θέλω σήμερα να σας ε, παρουσιάσω προέρχονται από μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Καταρχήν όμως θέλω να σας παρουσιάσω μια διαφάνεια που αφορά την περιοχή μου. Γιατί νομίζω ότι η μετάβαση στη, στον τομέα της ενέργειας πραγματικά είναι αποτέλεσμα της αποδοτικότητας ε, στον τομέα της ενέργειας και των ανανασιώσιμων πηγών. Βλέπετε εδώ την πρόοδο που έχουμε επιτύχει στην περιοχή μας, στη Βόρεια Αυστρία, Όμπερ Όστρια, και βλέπετε ότι πραγματικά κερδίζουν χώρο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην πάνω, στο πάνω μέρος αυτής της διαφάνειας βλέπετε το ποσοστό στο συνολικό ποσοστό ενέργειας. Είμαστε μια βιομηχανική περιοχή και βλέπετε τα ποσοστά όσον αφορά τη θέρμανση 61% και την βασική πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας 32%. Έχουμε βεβαίως και ενέργεια που προέρχεται από άλλες πηγές όπως την αιωλική ενέργεια, την ηλιακή ενέργεια. Αυτά όλα τα πετύχαμε τα τελευταία 10 χρόνια. Από το 2005 ως το 2015 μειώσαμε τις εκπομπές θερμοκηπίου κατά 43% και αυτό οφείλεται κυρίως σε πολύ αυστηρή, αν θέλετε, πολιτική για να αλλάξουμε το ενεργειακό μας μείγμα. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλες πηγές ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με έναν αποδοτικό και οικονομικό τρόπο. Είναι σαφές σήμερα ότι όταν κάποιος αρχίσει να αναφέρει τις νέες πηγές ενέργειας, αμέσως έρχεται το θέμα του κόστους. Όμως, όταν το ενεργειακό μείγμα αλλάζει ταυτόχρονα, η μετάβαση είναι πολύ πιο εύκολη και η συζήτηση λιγότερο έντονη. Βλέπουμε λοιπόν ότι το σχέδιο Energy Efficiency Watch, παρακολούθηση δηλαδή της αποδοτικότητας ενέργειας, είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 11.000 ε, εμπειρογνώμονες συμμετείχαν ε, απαντώντας σε ένα αριθματολόγιο. Αναλύσαμε τα δεδομένα. Πρόκειται για πραγματικούς ανθρώπους ε, επιτόπου οι οποίοι ουσιαστικά απάντησαν για το πώς αξιολογούν, πώς βλέπουν τις πολιτικές που εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη. Εδώ βλέπετε μία εικόνα Όσον αφορά τους δείκτες πρόοδου, δεν θέλω να, να κάνω κανένα σχόλιο όσον αφορά τις επιδόσεις των κρατών, αλλά βλέπετε την πρόοδο, τα βελάκια δηλαδή, προς τα πάνω ή προς τα κάτω οι αλλαγέ ε, κυβερνήσεων, η πολιτική λιτότητα παραδείγματος χάνει σε κάποιες χώρες, εξηγούν ε, ως ένα βαθμό αυτά τα βελάκια που ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν. Είναι λίγο ανησυχητικά βέβαια κάποια από αυτά που βλέπουμε. Σε κάθε περίπτωση οι πολιτικές παραμένουν φιλόδοξες και ένας από τους λόγους που βρήκαμε σαν απάντηση ε, γιατί αυτά τα προγράμματα υλοποιούνται, συνεχίζουν παρόλες τις ε, αντίξωες συνθήκες, είναι ότι πραγματικά δεν είναι κάτι που επιβάλλεται από τις Βρυξέλλες, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα πάνω, αλλά πραγματικά ο κόσμος θεωρεί ότι πρέπει αυτή η μετάβαση να γίνει. Βεβαίως υπάρχουν σοβαρές ε, διαφορές μεταξύ των χωρών. Υπάρχουν οι χώρες που στηρίζονται στην ε, ανεξαρτησία, που στηρίζονται σε κριτήρια όπως ε, κλιματική αλλαγή, ασφάλεια και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Βλέπουμε επίσης ότι εμείς οι εμπειρογνώμονες αλλά και οι πολιτικοί πρέπει να στηρίξουμε τις προσπάθειές μας σε ε, μια αφήγηση η οποία να περιγράφει όλα αυτά. Εδώ βλέπετε τώρα αυτές τις πολιτικές απόδοσεις σε σχέση με την αποτελεσματικότητά τους. Ποια είναι τα εργαλεία και τα μέσα που δουλεύουν στη χώρα σας, που είναι αποδοτικά στη χώρα σας. Αυτό που είναι εδώ εντυπωσιακό είναι ότι υπάρχουν εργαλεία που φαίνεται ότι σε κάποιες χώρες έχουν απόδοση είναι αποτελεσματικά σε όλες τις χώρες. Νέα κτίρια με νέο εξοπλισμό για ενεργειακή απόδειση. Όπως βλέπετε, ό,τι έχει σχέση με την κατασκευή κτιρίων είναι αποτελεσματικό. Με δύο λόγια, ρυθμιστικές, κανονιστικές διατάξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, μακροπρόθεσμες, και βεβαίως ε, αυτό είναι κάτι που ξεπερνάει τις αντικσότητες, Δηλαδή, λίγο πολύ οι ευρωπαϊκές οδηγίες είναι αυτές που κατευθύνουν και δίνουν την κατευθυντήρια γραμμή αυτών των πολιτικών που υλοποιούνται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στα κράτη-μέλη. Ένα στοιχείο που επίσης φάνηκε από, αυτή, την, ε, από αυτό το ερωτηματολόγιο είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερες επιχειρήσεις αυτό δεν είναι κάτι που περιμέναμε να το μάθουμε από το ερωτηματολόγιο, αλλά οπωσδήποτε κάποιες επιχειρήσεις αναπτύσσονται πολύ καλύτερα σε κάποιες χώρες και όχι σε άλλες. Και παραδείγματο χάρη είδαμε, εκεί που υπάρχει ένα οικονομικό πλαίσιο το οποίο επιτρέπει, διευκολύνει την ενεργειακή απόδοση σαν κύριο, αν θέλετε, αντικείμενο μιας επιχείρησης, σαν την καρδιά της οικονομικής δραστηριότητας, δείχνει ότι πολλαπλασιάζονται τα θετικά αποτελέσματα. Το άρθρο 7 της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση βλέπουμε ότι σε κάποιες χώρες εφαρμόζονται, σε άλλες όχι. Και το δυναμικό των χωρών αυτών σαφώς πολλαπλασιάζεται και με αυτόν τον τρόπο και άλλοι τομείς ανοίγουν στην ενεργειακή απόδοση βλέπετε πώς πλησιάζουμε αυτήν την πολιτική ενεργειακή απόδοσης. Είναι κάτι που θα πρέπει να συνδυάζεται βεβαίως και από κίνητρα αλλά και από κυρώσεις. Το καρότο και το μπαστούνι. Χρειάζεται μία αυστηρή ρύθμιση, ένα πλαίσιο, χρειάζονται κίνητρα οικονομικά, κίνητρα άλλου είδους, αλλά χρειάζεται βεβαίως να υπάρχει και μία αυστηρή παρακολούθηση της στήρησης. Και νομίζω ότι αυτό που σας είπα προηγουμένως, το αφήγημα είναι πολύ σημαντικό. Γιατί κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, υπάρχουν πολλοί άλλοι λόγοι. Συμπερασματικά, φιλόδοξοι στόχοι, πολιτικά μέτρα. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να υπάρχει διαλειτουργικότητα στα πολιτικά μέτρα που προτείνουμε και βεβαίως να πείσουμε και τους πολιτικούς αλλά και αυτούς που καλούνται να εφαρμόσουν αυτά τα πολιτικά μέτρα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ο τρίτος ομιλητής είναι ο James Drinkwater. Πίνει νερό ήδη. Φαντάζομαι ότι αυτό το αστείο θα το έχετε ακούσει πολλές φορές με το όνομά σας. Θα αναφερθούμε εδώ στις ε, περιφερειακές ε, στρατηγικές που θα μπορέσουν να συμπληρώσουν την γενικότερη ευρωπαϊκή στρατηγική. Ο κύριος Drinkwater είναι συντονιστής διαδικασιών παγκόσμιων και ευρωπαϊκών στον ε, χώρο της αηφόρου ανάπτυξης προγράμματα όπως το Horizon 2020 ε, με πάνω από 2.000 συμμετέχοντες από πολλές διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, στρατηγικές ανανέωσης σε εθνικό επίπεδο. Και στα πλαίσια του Horizon 2020 ε, προγράμματα που αφορούν την ενεργειακή απόδοση και προσφέρουν προγράμματα για τη βελτίωσή τους. Κύριε Drinkwater, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε, η οργάνωσή μου τα τελευταία δύο χρόνια συντώνησε αυτή τη τεράστια προσπάθεια που εστιάζει στο σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων πολιτικών. Οργανώσαμε 100 εκδηλώσεις σε όλα τα κράτη-μέλη, στις μεγαλύτερες πόλεις αυτών των κρατών και χαίρομαι πολύ που έχω την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας κάποια διδάγματα. Οι στρατηγικές ε, ανακαίνησεις συμβάλλουν ε, στην ανάπτυξη της ε, οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση. Η πρόκληση της ανακαίνιση είναι πολύπλοκη. Υπάρχουν πολίτες στη καρδιά ε, των πολιτικών που εφαρμόζουμε, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και άλλο να έχουμε να κάνουμε με ε, ε, οργανισμούς και άλλο με ε, πέτρες. Όταν έχουμε να κάνουμε με ένα ζωντανό πολύπλοκο οργανισμό όπως ένα πουλί, δεν μπορούμε να προβλέψουμε ακριβώς τη διαδρομή που θα φτάσει. Ένα από τα σημαντικότερα διδάγματα λοιπόν είναι να σταματήσουμε να προσπαθούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο και να σχεδιάσουμε ε, αποτελεσματικές στρατηγικές. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να σας πω είναι ότι η δημόσια διαβούλευση είναι κλειδί σε μια επιτυχημένη στρατηγική ανακαίνιση. Χτίζουμε, ξεκινήσαμε να χτίζουμε, να οικοδομούμε πλατφόρμες σε κάθε κράτος μέλος όπου δραστηριοποιούμαστε. Μιλήσαμε για μετρήσεις, ε, αξιολογήσαμε την ποιότητα της ε, συνεργασίας και των δεσμεύσεων προκειμένου να συνεργάζονται οι κατάλληλοι παράγοντες. Και μπορώ να σας πω ότι οι παράγοντες της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν συνεργάζονται πάντα με τον βέλτιστο τρόπο. Πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε και στον σωστό σχεδιασμό σε ε, κοινοτικό επίπεδο αυτό είναι πολύ σημαντικό για να ε, ενώσουν τις δυνάμεις τους όλες οι ομάδες ε, φορέων και παραγόντων. Γιατί κάτι τέτοιο θα ορίσει και την ποιότητα της λύσης. Είναι πολύ σημαντική η προσέγγιση που θα ακολουθήσουμε. Στο παρελθόν ποτέ δεν συνεργάστηκαν ε, τράπεζες, παράγοντες του τομέα της ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του τομέα των κατασκευών. Αυτό όμως πετύχαμε αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι κλειδί και πρέπει να ενισχύσουμε μια τέτοια προσέγγιση. Δεύτερον, πρέπει να περάσουμε στο συντονισμό συλλογικών πλαισίων στις οργανώσεις σας θα ε, προσλαμβάνατε 100 άτομα χωρίς να έχετε την απέτηση να λογοδοτούν. Εμείς ανακαλύψαμε ότι ε, σε κάθε κράτος μέλους υπάρχουν ε, πολλά έργα σύμπραξης ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, στον τομέα της ανακαίνησης, που ε, εστιάζουν στη χρηματοδότηση, την ευαισθητοποίηση του κοινού μεταξύ άλλων και ε, συμπεράνουμε ότι πολύ μικρό ποσοστό αυτών των ε, πρωτοβουλειών δημοσιεύουν τα αποτελέσματα και την πρόοδο. Χρησιμοποιείται λοιπόν τεράστια ποιότητα, ε, ε, ποσότητα πόρων, αλλά δεν ε, δίνονται αναφορές για τα αποτελέσματα. στο τομέα των χρηματοδοτήσεων, της ευαισθητοποίησης, των δεξιοτήτων. Όλοι αυτοί οι τομείς άρχισαν να συνεργάζονται, να δουν ποιοι μπορεί να είναι οι κοινοί στόχοι, γιατί μέχρι τώρα ακολουθούσαν διαφορετικούς δρόμους χωρίς να γνωρίζουν ότι υπάρχουν κοινοί στόχοι και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να έχουμε τις αποτελεσματικότερες ε, λύσεις. Είναι σημαντικό να συνεργαστούν όλοι οι τομείς. Φανταστείτε μία εταιρεία κατασκευών σημαντικό κομμάτι της δουλειά θα το κάνει ε, μία ομάδα μηχανικών, αλλά υπάρχουν και άλλα τμήματα ε, σε αυτή την επιχείρηση που θα συμβάλλουν, όπως το τμήμα marketing. Είναι σημαντικός ο συντονισμός της ομάδας. Και, κάτι άλλο που θα ήθελα να πω, σε ό,τι αφορά τα ενυπόθηκα δάνεια για την ενεργειακή απόδοση, είδαμε ότι για κάθε κτίριο είναι σημαντικό να έχουμε στόχο την μηδενική ενεργειακή κατανάλωση. Και πρέπει να το έχουν υπόψη τους αυτό οι επενδυτές. Πρέπει να βεβαιωθούν ότι τα κτίρια είναι ανθεκτικά και να υπάρχουν μακροπρόθεσμα σχέδια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να ε, γίνει ο κατάλληλος σχεδιασμός για κάθε κτίριο ως προς την ε, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, προκειμένου οι επενδυτές να αρχίσουν να χρηματοδοτούν την ανακαίνιση των εν λόγω κτίριων. Τέλος θα ήθελα να σας επανέλθω στο θέμα των ανθρώπων. Μιλάμε για την οικονομική απόδοση της ανακαίνεσης των κτηρίων με τις κατάλληλες προσεγγίσεις και τη χρήση, τη χρήση ανανεμώσιμων πηγών ενέργειας. Μιλάμε για τον κανόνα των 90 σε ένα κτίριο με γραφεία. Δεν πρέπει να βασιστούμε στο κόστος της ενέργειας. Ε, κλειδί είναι οι ανθρώπινοι πόροι. Και ο υπεύθυνο των οικονομικών θεμάτων ενδιαφέρεται για την, ε, τη σχέση ανάμεσα στην απόδοση των ανθρώπων και την ενεργειακή απόδοση. Πρόκειται για πολύ σημαντικό τομέα στον, οποίο υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Πρέπει να επενδύσουμε σε εργαλεία που θα ε, βασίζονται στην ε, συσχέτιση της μέτρησης των περιβαλλοντικών παραγόντων και της ενεργειακής ε, απόδοσης. Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια έρευνα σε αυτό το τομέα. Μίλησα για την στρατηγική ανακαίνησης και κλείνοντας θα ήθελα να κλείσω με ένα πιο αισιόδοξο μήνυμα Νομίζω ότι είναι σημαντικό να συνεργαστούν όλοι, ε, όλοι οι παράγοντες σε ένα κοινό ε, ταξίδι. to... Κύριε Drinkwater, σε ευχαριστώ πολύ. Το παράδειγμα που δώσατε με το πουλί και την πέτρα μου θύμιζε αυτό που όταν δούλευα σε μια αμερικάνικη εταιρεία έλεγαν ότι δεν τους φοβόμαστε τις άγριες πάπιες όσο πετάνε σε σχεδιασμό. Ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις οικοδομές. Ο κ. Βάουτερ είναι ε, Διευθυντής Ανάπτυξης και Αξιοποίησης στο Ινστιτούτο Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας του Βελγίου. ποιοτικές βελτιώσεις στον τομέα των οικοδομών και ε, ο ρόλος των ρυθμιστικών αρχών στις τεχνικές βελτιώσεις και τις αξιολογήσεις. Κύριε Βάουτερς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τρία συμπεράσματα, τα οποία θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω εκ των υστέρων. Καταρχάς, οι υπεύθυνοι για την πολιτική και το σχοδιασμό και εφαρμογή των πολιτικών θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη διευκόλυνση της αξιολόγησης των καινοτόμων τεχνολογιών και των ελεγκτικών τεχνολογιών. Ε, η κατασκευή των κτηρίων θα πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε μια ευφυή εφαρμογή των ενεργειακών πολιτικών, κάτι το οποίο απαιτεί προετοιμασία εκ των προτέρων. Οι πολιτικές ανακαίνισεις και οι λύσεις που βρίσκονται δεν θα πρέπει να παραμένουν μόνο στις σημερινές λύσεις, αλλά να φέρονται και σε μελλοντικές δυνατότητες. θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε τις πολιτικές αυτές όχι μόνο στα νέα κτίρια αλλά και στα υπάρχοντα κτίρια. Οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές, είναι προκλήσεις πολλές που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ε, του συνόλου των κτιρίων που υπάρχουν σήμερα θα πρέπει να μειωθεί μέχρι το 2050, κάτι το οποίο είναι προβληματικό οικονομικά το τεχνολογικό πλαίσιο τώρα έχουν ε, υπάρξει ενδιαφέρουσες εξελίξεις στον τομέα της οικοδομής και στον τομέα των συστημάτων και των συστημάτων ελέγχου και ακούσαμε ότι μέχρι το 2050 τα ανανεώσιμα θα καλύψουν μεγαλύτερα ποσοστά αναγκών. Ας δούμε τώρα τα υλικά συστήματα και τα νέα υλικά που χρησιμοποιούνται. Βλέπουμε να υπάρχουν πολλές βελτιώσεις. Μερικές φορές είναι ριζοσπαστικές οι αλλαγές οι οποίες υπάρχουν. Αν δει κανεί τις ε, εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν στον τομέα των ανανεώσιμων, θα δει ότι υπάρχουν και εντελώς νέα συστήματα που χρησιμοποιούνται και υπάρχουν και ευφυείς τεχνολογίες με πάρα πολύ υψηλό δυναμικό. Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν την δυνατότητα να καλύψουν τη ζήτηση της ενέργειας, υπάρχουν δυνατότητες για βελτίωση της αποτελεσματικότητας της παραγωγής ενέργειας, κάτι το οποίο θα είναι χρήσιμο για τους πολίτες. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις επίσης σε μεμονωμένα κράτη-μέλη. Τα θέματα των εθνικών νομοθετικών ρυθμίσεων θα πρέπει να αντιμετωπιστούν έτσι ώστε όλες αυτές οι καινοτόμες τεχνολογίες να λαμβάνονται υπόψη στους εθνικούς υπολογισμούς. Αλλιώς μπορεί να υπάρξει μια διασπορά η οποία δεν θα βοηθήσει το ολοκληρωμένο του συστήματος. Εμείς έχουμε προχωρήσει με το λεγόμενο πρόγραμμα QualiCheck, το οποίο δείχνει ότι σε πολλές χώρες υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα χρήσης των καινοτομιών, στην ουσία λειτουργούμε σαν τροχοπέδι για τις ε, τεχνολογίες αυτές. Τώρα για τις κατασκευές 4.0 και BIM ξέρετε ότι χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο τα drones, τα μη επανδρομένα πτήτικα συστήματα για την διαδικασία σχεδιασμού και ελέγχου της οικοδομικής δραστηριότητας. Νομίζω ότι ήταν το BIM, το BIM, κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν βέβαια αρκετές δυσκολίες οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν. Είναι σαφές ότι όταν προχωράμε προς το NZEB θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αυξημένη περιπλοκότητα την οποία επιβάλλουν οι νέες μορφές σχεδιασμού εκτεκτονικής η μεταφορά των κανόνων των νέων μερικές φορές λειτουργεί σαν τροχοπέδι στην καινοτομία. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία είναι δύσκολο να αντιμεταπιστούν όπως η υπερθέρμανση μηχανισμών. Βλέπουμε να υπάρχει περιορισμένη συμμόρφωση από τους ελέγχους ή από τις προσπάθειες τις οποίες κάνουμε επιβολής κανόνων. Βλέπουμε επίσης ότι αν ε, και υπάρχουν ομοιότητες ε, στους στόχους ανάμεσα στις χώρες, είναι δύσκολο να ελέγξουμε από κοινού τους τρόπους με τους οποίους ακολουθούν οι χώρες για να το πετύχουν. είναι επίσης αρκετά δύσκολο να έχουμε μια ευφυή αξιολόγηση της έννοιας της ευφυΐας στην οικοδόμηση. και να δούμε ακριβώς το πώς θα αξιολογήσουμε καλύτερα τις ανανεώσιμες πηγές όχι μόνο στην φάση της οικοδομής αλλά και σε γενικότερα κοινωνικό επίπεδο. Τώρα το BIM και το 4.0 ε, πρέπει να υπάρξουν βελτιωμένες προσπάθειες συλλογής δεδομένων. Θα πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα όχι μόνο για την ενέργεια αλλά και για τα υπόλοιπα στοιχεία ενδιαφέροντος. Θα πρέπει να απλοποιήσουμε το πλαίσιο αυτό και να προχωρήσουμε σε πιο εκλεπτισμένες μορφές ανάλυσης. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο για τις δυνατότητες συμμόρφωσης θα πρέπει επίσης να καταστήσουμε τον σχεδιασμό ε, πιο, ε, θα έλεγα, ανοιχτό στην καινοτομία, να αυξήσουμε τις δυνατότητες μιας πραγματικά ευρωπαϊκής μεθόδου IPBD e και να ε, βελτιώσουμε την ποιότητα των εργασιών και νομίζω ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε μεγαλύτερο χώρο για την σωστή περιβαλλοντική αξιολόγηση του BIM. Έτσι λοιπόν υπάρχει ανάγκη για τις ρυθμιστικές αρχές να δούνε με ποιο τρόπο θα εντάξουν το BIM και θα πρέπει να υπάρξει και προσπάθεια επίσης βελτιστοποίησης των επιπέδων τα οποία θα πρέπει να γίνονται γενικώ παραδεκτά και σεβαστά. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ακριβώς και το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την εφαρμογή των ανανεώσιμων Νομίζω ότι αν δούμε το 2050 με τις σημερινές λύσεις δεν επαρκεί, θα πρέπει να βελτιώσουμε στην πόλη αυτή σαν παράδειγμα πολύ καλύτερα την μόνωση στα κτίρια παλαιά και νέα. Θα πρέπει να υπάρχουν ε, boilers πύκνωσης, τα οποία μπορεί να είναι μια καλή επιλογή, αλλά σε 20 χρόνια θα είναι ανάγκη, θα έλεγα, να χρησιμοποιούμε άλλα προϊόντα για θέρμανση, όχι φυσικό αέριο ή άλλα καύσιμα ορυκτά, οπότε δεν θα έχουμε ανάγκη πλέον τα boilers. Δεν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τις περιφερειακές μορφές θέρμανσης και ψήξης, όπως επίσης και τους θερμοπομπούς. Να ελέγξουμε το πόσο λοιπόν μονομένα και σωστά μονομένα και αεροστεγή είναι τα ακτήρια να μην δημιουργούμε ή μάλλον να δημιουργούμε ε, κενά στις, στους φέροντες τείχους οι οποίοι να μην είναι μονομένοι γιατί η μόνωση αυτή στο εσωτερικό των τείχων είναι κάτι το οποίο κοστίζει και θα πρέπει επίσης να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και σε σχέση με τη μόνωση των δαπέδων στα νέα κτίρια. Λοιπόν, αυτά ήταν γενικά τα συμπεράσματα τα οποία ήδη σας παρουσίασα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Φορετικούς τρόπους ε, ε ασφαλούς χρήσης της ε, ηλεκτρικής Είναι επίσης πρόεδρος της Ισπανικής Οργάνωσης ε, Θέρμανσης και Ψήξης. Έχετε το λόγο. Η παρουσίασή μου θα γίνει στα Ισπανικά. Eh, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Είναι θετικό για μας ε, το ότι βρισκόμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε τις εμπειρίες μας, ιδιαίτερα σε σχέση με τη χρήση συγκεκριμένων μεθόδων όπως τα φωτοβολταϊκά. να πω ότι η περιοχή μας βρίσκεται στα νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας, της Ισπανίας και της Ευρώπης. Είναι σημαντικές οι ανανεώσιμες πηγές, έχουμε και υδροηλεκτρική ενέργεια, αλλά κυρίως έχουμε ηλιακή ενέργεια. Βλέπουμε ότι έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της χρήσης φωτοβολταϊκών και αυξάνεται συνεχώς η χρήση τους να σας μεταφέρω κάποια δεδομένα τα οποία γνωρίζετε ίσως τη σημασία που έχει δηλαδή ε, η χρήση των φωτοβολταϊκών. Έχει αυξηθεί επαναλαμβάνω τα τελευταία χρόνια 105% την τελευταία δεκαετία έχουν επίσης βελτιωθεί οι διάφορες μορφές αποδοτικότητας της συγκεκριμένης ενέργειας δεν απαιτούνται σημαντικές τεχνολογικές εγκαταστάσεις. Το ηλεκτρικό δίκτυο κερδίζει λοιπόν σε επίπεδο αποδοτικότητας κατά υψηλότατα ποσοστά που φτάνουν μερικές φορές και το 70%. Αυτό το σημαίνει ότι δεν δημιουργούνται περιβαλλοντικές επιπτώσεις μέσω της χρήσης των φωτοβολτιακών στις κατοικίες. Αποφεύγουμε λοιπόν συνέπειες στον τομέα της, του περιβάλλοντος. Και ένα τελευταίο στοιχείο είναι ότι μειώνουμε και τις εκπομπές κατά 40% συνολικά και έχουμε μειώσει ήδη τις εκπομπές σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και αυτό οφείλεται ακριβώς ε, στην χρήση των φωτοβολταϊκών. Θα μπορούσαμε να καλύψουμε το 80% των κατοικιών σε επίπεδο ενέργειας μέσω ακριβώς της χρήσης των φωτοβολτιακών σε πολλές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, υπάρχει όμως μια κάποια θα έλεγα αστάθεια σε σχέση με τις νομικές ρυθμίσεις οι οποίες καλύπτουν ε, τον τομέα αυτό. Πάντως ε, το, η ζήτηση στην περιοχή μου είναι ιδιαίτερα υψηλή σε Ιταλία, Ελλάδα καλύπτουν το 5 με 7% και ταυτόχρονα σε χώρες όπως ε, η Δανία το ποσοστό αυτό ε, καλύπτεται σε διπλάσιο ποσοστό από ότι ε, στην Ισπανία. Το κόστος βέβαια των εγκαταστάσεων στις χώρες αυτές είναι υψηλότερο, αλλά παρόλα αυτά στην Ισπανία υπάρχουν συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις, στην Εστρεμαδούρα σαν παράδειγμα προβλέπεται να υπάρχουν οικονομικά βοηθήματα που καλύπτουν το 20 με 40% του κόστους εγκατάστασης. Έχουμε 1,5 λοιπόν μεγαβάτ παραγωγής άμεσης κατανάλωσης και έχουμε επίσης και δυνατότητα συσσωρευτών σε περιορισμένο προς το παρόν επίπεδο. Εδώ βλέπετε πόση δημολογήσεων και τέλος υπάρχει και ε, δυνατότητα πληρωμής για την ενέργεια η οποία παράγεται σε οικιακό επίπεδο φωτοβολταϊκών στην αυτοκατανάλωση και βλέπουμε και στα κίτρινα Τσεχία, Πορτογαλία, Μάλτα, Σουηδία κτλ. Ε, και υπάρχουν σημαντικές διαφορές βέβαια στις νομοθετικές δραστηριότητες οι οποίες όμως ισχύουν ε, σε κάθε δύο με τρία χρόνια αλλά υπάρχουν μερικές φορές καθυστερήσεις και στρεβλώσεις. Το πρώτο παράδειγμα Έχουμε και διαφορετικά παραδείγματα τα οποία οδηγούν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Βλέπουμε μια εγκατάσταση σαν παράδειγμα στην Ισπανία, κάτι το οποίο χρησιμοποιούν τα φωτοβολταϊκά. Βλέπουμε ακριβώς τι γίνεται στη Γερμανία. Υπάρχει μια αρχική ε, επένδυση. Πάρα πολύ σύντομα λοιπόν Βλέπουμε ότι θα πρωταγωνιστήσουν τα φωτοβολταϊκά και τέτοιου είδους μορφές παραγωγής ε, ηλεκτρικής ενέργειας ε, στο μέλλον. Αλλά θα πρέπει συνεχώς ε, το θεσμικό πλαίσιο το θέμα είναι να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας επίσης ανάμεσα σε διαφορετικές περιοχές και και βλέπουμε ότι θα μπορούσε να... Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα είδος κινήτρων. Υπάρχει η δυνατότητα, αν θέλετε, εφαρμογή σε κάποιον. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τις δυνατότητες αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Και προτείνεται επίσης και ε, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρξουν δυνατότητες με καταπιστεύματα εγγυήσεων. Δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε τις νέες τεχνολογικές λύσεις που διαθέτουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο Τόμας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις ε, εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και υψηλού επίπεδου παρουσιάσεις. Μιλήσατε για τα νέα κτίρια, για τον κατασκευαστικό τομέα. Εκεί τα πράγματα είναι πιο εύκολα όσον αφορά τον εξοπλισμό, αλλά το πραγματικό... Και εκεί υπάρχουν πολλές διαφορετικές δυσκολίες, όπως παρουσιάζουν η υπεύθυνη του κατασκευαστικού τομέα. Πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα ακούγοντάς, σας, ακούγοντάς να μας λέτε στον τομέα αυτό. Το θέμα της ε, ανακαίνησης των κτηρίων. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα είδους ε, πιστοποίησης. Χρειάζεται μία ανακαίνιση η οποία να γίνεται σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε μία εβδομάδα παραδείγματος χάρη και όχι σε οχτώ μήνες. Και βεβαίως θα πρέπει να δούμε και τις οικονομικές συνέπειες. Σήμερα μπαίνουμε, λοιπόν, πολύ σημαντικό να ξαναδούμε την ανακαίνιση όλων αυτών των κτίριων και να είναι αερίων του θερμοκηπίου Κηπίου. Δεν μπορεί να αφήνουμε τον ιδιοκτήτη να παίρνει αποφάσεις για την ανακαίνιση. Αυτό θα πρέπει να γίνεται συνολικά. Έχετε τέτοιο για την ανασυνεώσιμη πηγή ενέργεια του 34%. Δηλαδή είναι κάτι που επανήλθε. Αυτό που με... Πραγματικά σήμερα δείχνουν ε, σημαντικές ε, προσπάθειες και βούληση για μία παραγωγή χωρίς άνθρακα, με χρήση νέων τεχνολογιών. Και αυτό βεβαίως σε όλους τους να συνειδητοποιήσει ότι σε όλους τους τομείς ε, ο περιορισμός του άνθρακα είναι σήμερα το ζητούμενο. Και στα κράτη-μέλη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία, αυτή την τάση βλέπουμε νέους κατασκευές χωρίς να προβλέπεται ο εξοπλισμός τουλάχιστον λοιπόν στα νέα κτίρια θα πρέπει να αναφορά την το κατανάλωση. Οι περισσότεροι καταναλωτές δεν γνωρίζουν τις δυνατότητες που υπάρχουν. Δεν ξέρουν ακριβώς ε, πώς θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν με αποτελεσματικό τρόπο ενέργεια και δράσουν μηνύματα και εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να βοηθήσουμε και να περάσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρούμε ότι και η εθνική και η ευρωπαϊκή ε, τις διαφορές ε, που υπάρχουν οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική ανάπτυξη. Και μιλήσατε λοιπόν για τα πουλιά. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πουλί σε κλουβί. Ένα μεγάλο ποσοστό των κτηρίων, πολύ σημαντικά κτίρια στις πόλεις μας, ανήκουν στις κυβερνήσεις, πρμίσουν και να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση αυτών των κτίριων. Μία απλή ερώτηση που αφορά γραφεία σε δημόσια κτίρια, σε βιομηχανικά κτίρια και για κατοικίες. Κύριε Καθηγητή, πιεστική. Φυσικά Καταρχήν θα σας δώσω το λόγο να απαντήσετε, αλλά αν υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις θα υπάρξει και ένας δεύτερος γύρος, αν έχουμε χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Να απαντήσω καταρχήν στο αν πρέπει η στόχη να είναι εθνική ή ευρωπαϊκή. Φαντάζομαι αναφέρεστε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. για το 2020 υπάρχουν και ευρωπαϊκοί και εθνικοί στόχοι και είναι κρίμα πραγματικά που αυτό δεν έχει τεθεί και για το 2030. Ο βασικός λόγος είναι ότι δημιουργείται μία αβεβαιότητα για τους επενδυτές. Πιστεύω ότι οποιοδήποτε και να είναι ο στόχος που τελικά θα αποφασιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το 2030 θα πρέπει να οδηγήσει όλες τις χώρες να προσαρμοστούν σε αυτό. Αυτό δεν είναι βέβαια ιδανικό, αλλά ελπίζω να οδηγηθούμε σε περισσότερη σαφήνεια με αυτόν τον τρόπο όταν αποφασιστούν οι στόχοι. Στη δεύτερη ερώτησή σας, ε, βεβαίως και έχουμε την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά έχουμε και το διοξίδιο του άνθρακος, έχουμε και τις εκπομπές ε, του θερμοκηπίου και εννοείται ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε πως η ενεργειακή πολιτική σαφώς και ενδυναμώνει τους υπόλοιπους τομείς ε, πολιτικών και αποφάσεων επίπεδο, σίγουρα αποτελούν μια, έναν σταθεροποιητικό παράγοντα για τις υπόλοιπες αποφάσεις. Κυρία Έγκερς, ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω με την ερώτηση του κυρίου Τούρμες. Αυτό που πραγματικά θα θέλαμε και θα βοηθούσε πάρα πολύ τη δική μας προσπάθεια είναι να απαγορευθούν οι καυστήρες πετρελαίου στα νέα κτίρια. Πιο αυστηρές δηλαδή ρυθμίσεις. Εάν τουλάχιστον στα νέα νομοθετικά πλαίσια υπάρχουν κίνητρα δεν μπορείτε να επιβάλλετε κάτι, αλλά να δώσετε κίνητρα στα κράτη-μέλη τουλάχιστον να απαγορεύσουν αυτού του είδους τους ε, ε, καυστήρες στα νέα κτίρια. Νομίζω, νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει πολύ. Τουλάχιστον δηλαδή θέτουμε ένα πλαίσιο νομοθετικό για τις κυβερνήσεις αυτές που θέλουν να είναι φιλόδοξες. Εγώ σήμερα είμαι επικεφαλής στη χώρα μου σε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία στον τομέα της βιομηχανίας, της κατασκευαστικής, ε, του κατασκευαστικού τομέα. Και το κύριο μήνυμά μας είναι ότι η μείωση περιεκτικότητας σε άνθρακα σε όλους αυτούς τους τομείς, μακροπρόθεσμα, δεν αποτελεί εμπόδιο, αλλά αντίθετα διευκολύνει την βιομηχανική παραγωγή και πιστεύω ότι οι στόχοι, και εδώ απαντώ στην άλλη σας ερώτηση, θα πρέπει να είναι σε όλα τα επίπεδα, και τοπική, και περιφερειακή, και εθνική, και ευρωπαϊκή. Μιλήσατε για το πώς αξιολογούμε την ε, απόδοση των κρατών, ότι έχουμε κάνει ένα είδος ε, καταλόγου, πίνακα αξιολόγησης. Δεν θελήσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, να βάλουμε βαθμολογίες. Αλλά αυτά τα αποτελέσματα που σας έδειξα είναι πραγματικά πώς αξιολογούν οι εμπειρογνώμονες τα προγράμματα και τις πολιτικές που υλοποιούνται στις διάφορες χώρες μέλη μετά τα και θα πρέπει να μην υπάρχει γραφειοκρατία η οποία να επιβαρύνει τη διαδικασία αυτή και να την κάνει μη ελκυστική. Και θα πρέπει να μην υπάρχει γραφειοκρατία η οποία να επιβαρύνει τη διαδικασία αυτή και να την κάνει μη ελκυστική. Υπάρχουν οι διαδικασίες για να γίνουν πιο δημοφιλή αυτά τα δάνεια. Μιλήσατε για τα δημόσια κτίρια. Μία παραδειγματική, αν θέλετε, διαδικασία ανακαινήσεων. Αλλά βεβαίως αυτό δεν γίνεται ούτε σε όλες τις χώρες και... μέσω των κατασκευών πρέπει να επενδύσει στις δεξιότητες να γίνουν κατάλληλες πρωτοβουλίες. Συμμετείχα τη Δευτέρα σε μία κατασκευών. Πρέπει να γίνουν πιο αποτελεσματικές Ο τομέας γνωρίζει τις προκλήσεις και στο μέλλον θα υπάρξουν βελτιώσεις. Και το θέμα της δεν θα συμβάλλει στο θέμα των δεξιοτήτων και στη βελτίωσή τους και αυτό θα, ε, θα απαντήσει ότι υπάρχουν ε, διαφορές ε, Σήμερα όμως πιστεύω ότι είναι καλύτερη μια πιο γενική Όποιο και αν είναι το είδος του κτηρίου, ε, πρέπει να ακολουθήσουμε την ίδια προσέγγιση. Χρειάζεται μια ολική προσέγγιση. Κύριε η επίδραση, το πόσο αλληλένδετες είναι η ενεργειακή απόδοση και οι ανανεώσιμες πηγές ε, ενέργειας πώς τοποθετήστε όσον αφορά το θέμα των τομέων αυτών, πολλοί τομείς όπως το κινητοβιομηχανία που συνεχίζουν να, να χρησιμοποιούν παραδοσιακές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βεβαίως υπάρχει βούληση να πάμε προς τα εκεί, αλλά δεν είδα να υπάρχει και μεγάλος ενθουσιασμός από όλα τα μέρη δεν πιστεύετε ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει πιο πιεστική, να γίνουν δεσμευτικοί οι στόχοι αλέξουν μόνο οι πλούσιες χώρες. Πώς βλέπετε λοιπόν όλα αυτά τα θέματα των ενεργειακών επιλογών στις φτωχότερες ε, χώρες, στις χώρες με προβλήματα ανάπτυξης. Χωρίς ενεργειακή απόδοση, πολλά κτίρια για την ενεργειακή απόδοση. Τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη και ο δυτικός κόσμος ε, γι' αυτό. Νομίζω ότι υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις, τις γνωρίζουμε και θα πρέπει κάποιος να τις επιβάλλει. Ο κύριος Τούρμες. Θέλω να συνεχίσω σε αυτό. Εχθές μιλήσαμε για το θέμα των δεξιοτήτων. Είχα μια συνάντηση χτες με την περιοχή στη Γαλλία του Λίγυρα. Υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα και εθνικά προγράμματα θεωρείτε ότι αυτά θα παραμείνουν ε, καθαρά τοπικά αυτά τα θέματα, ότι δηλαδή ο κατασκευαστικός τομέας από μόνος του δεν μπορεί παρά να είναι αρμοδιότητα των περιφερειών ε, τοπική, σε τοπικό επίπεδο. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις δεξιότητες σε τοπικό επίπεδο στον τομέα αυτόν. Υπάρχει και ένα λόμπι, αν θέλετε, για το οποίο τις ε, προσπάθειες να βελτιώσουμε τα κτίρια, την απόδοσή τους ε, όσον αφορά την ενέργεια, αντισταθούμε σε αυτό το λόμπι. Ποια είναι η εμπειρία σας. Πρέπει κάπως να σταματήσουμε να είμαστε αφελείς. Τον που ήθελα να κάνουν ερωτήσεις. Ποιος ε, θέλει να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις που έγιναν. Δεν θα απαντήσω εγώ, δεν θα αποφασίσω εγώ. Um, Σχολιάζοντας και τις δύο ερωτήσεις, ή μάλλον στη γερμανική. member states τα κράτη-μέλη μπλοκάρουν ουσιαστικά κάποιες υποθέσεις τις οποίες ε, οι τοπικές αρχές και οι περιφερειακές αρχές αντίθετα θέλουν να προωθήσουν. Αυτό δεν είναι κάτι το καινούριο. Το θέμα είναι να βλέπει κανείς σε τοπικό επίπεδο το τι έχει αξία. Εμείς έχουμε αγκυρώσει τις πολιτικές μας στην προστασία, αν θα έλεγα, από τις κλιματολογικές αλλαγές. Αν όμως προσθέσουμε επιχειρήματα όπως η ανταγωνιστικότητα, σαν παράδειγμα, στη χώρα μου υπήρξε αλλαγή κυβέρνησης και όλες οι πολιτικές ασχολούνται με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και στην ουσία παραμένουν ε, τα προβλήματα όσοι είχαμε. Από την άλλη εμφανίζονται θέματα για συζήτηση τα οποία η κυβέρνηση στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι διατεθειμένη να προωθήσει. Αυτό το οποίο ισχύει λοιπόν για τα κράτη-μέλη είναι κάτι το οποίο μπορεί να ισχύσει για όλους όσους διστάζουν μεταξύ των οποίων και για τους ιδιοκτήτες ε, κατοικιών. Λοιπόν, θα πρέπει να πετύχουμε ακριβώς το τι τους ευαισθητοποιεί. Σαν παράδειγμα, ένα κίνητρο θα μπορούσε να είναι η αύξηση της αξίας των ε, ιδιοκτήσεών τους. Και η κατασκευαστική βιομηχανία στη δική μου περιοχή είναι τοπική. Τοπική, τοπική, ούτε καν περιφερειακή, πόσο μάλλον όχι εθνική. Συνεπώς λοιπόν απασχολούνται άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την Αυστρία, δεν ομιλούν τη γερμανική και το θέμα είναι ότι αν ο πελάτης επιμένει τότε ανταποκρίνεται. Βλέπουμε ας πούμε ότι ε, οι επιχειρηματίες προσπαθούν να αποτρέψουν ε, τους ε, ιδιοκτήτες να χρησιμοποιήσουν φωτοβολταϊκά. Αλλά από την άλλη όταν επιμένει ο ιδιοκτήτης νομίζω ότι με τη βοήθεια και από την εθνική διοίκηση μπορεί να υπάρξει. Ο κύριος Βάουτευς κλείνοντας τη συζήτηση. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Νομίζω ότι οι ικανότητες στον τομέα της οικοδομής είναι τοπικές. Αλλά νομίζω ότι και ο ρόλος της Ευρώπης μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικός. Είχαμε ξεκινήσει μια προσπάθεια για την ομογενοποίηση των απαιτήσεων στον τομέα. Συμβαίνει στις διάφορες χώρες. υπάρχουν μέσα τα οποία είναι χρήσιμα για διαφορετικές χώρες ταυτόχρονα. Έχω την αίσθηση ότι το θέμα είναι εθνικό, αλλά υπάρχει και ξεκάθαρη δυνατότητα παρέμβασης για κινητοποίηση των δραστηριοτήτων. Για τις διάφορες χώρες πράγματι υπάρχει εδώ ένα κενό στον τομέα των γνώσεων έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και στις τεχνολογίες και δεν είναι όλοι ενήλικοι ένα ανανεώσιμων, έχει μακροοικονομικές συνέπειες θεπικές δημιουργεί θέσεις στην Ευρώπη και βοηθά το εμπορικό ισοζύγιο της Ευρώπης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο απαιτεί περισσότερη προσοχή. Σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήταν καλό να υπήρχε μια τιμή σαν παράδειγμα για το διοξίδιο που με συζητήσει εμείς και σε επίπεδο αποδοτικότητας και ανανεώσιμων αλλά και υψηλότερης άνεσης για τους ανθρώπους οι οποίοι κατοικούν στα κτίρια αυτά. Και ένα τελικό ε, σημείο, υπάρχει ένα πρόγραμμα στην Ολλανδία, ε, το οποίο σοπούν ακριβώς τα λόμπι αυτά για να δούμε τι ε, θα μας απαντήσουν. Σας ευχαριστώ όλους για τις εξαιρετικές σας παρουσιάσεις και τώρα θα δω... Uh, Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, ας ξεκινήσουμε χωρίς καθυστέρηση, να μην χάσουμε άλλο χρόνο. Το θέμα είναι πάρα πολύ γνωστό. Σας καλημερίζω και από πλευράς μου όλους. Συγγνώμη, αλλά δεν ήμουν διαθέσιμος ε, ε, στο hearing που προηγήθηκε. Αναγκαζόμαστε να είμαστε ταυτόχρονα σε πάρα πολλά μέρη και ήταν δύσκολο για μένα να είμαι εδώ παρόν. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τον επόμενο τριμερή διάλογο πάρα πολύ γρήγορα, σύντομα, για τα ανανεώσιμες. Χθε συναντηθήκαμε με εκπροσώπους των κυβερνήσεων, Νομίζω ότι ξεκινήσαμε με αρκετά επιτυχημένο τρόπο σε συνεργασία με την Επιτροπή ΕΝΒΗ. Βρισκόμαστε λοιπόν εν μέσω μιας μεγάλης μάχης για το πακέτο πράσινης ενέργειας και σας είμαι ευγνώμων που πήρατε όλοι μέρος στις συζητήσεις μας μέχρι τώρα. Έχει σημασία τέτοιου είδους ε, ακροάσεις, έχουν μεγάλη σημασία για τα ανανεώσιμα και την αποδοτικότητα. Χθε, όπως ενθυμίστε επίσης, είχαμε και μία ακρόαση για την εσωτερική αγορά στον τομέα του φυσικού αερίου και σήμερα θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά στον τομέα του φυσικού αερίου. Δεν νομίζω ότι πρόκειται να περάσω σε τεχνικά θέματα. Υπάρχουν 142 τροπολογίες, δεν είναι πάρα πολλές. Πρόκειται για μια πάρα πολύ σύντομη οδηγία τριών σελίδων, ίσως είναι η πιο σύντομη που έχω συναντήσει, δεν είναι πολύ περίπλοκη η κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ουσία προτείνει την αναθεώρηση της ισχύουσας οδηγίας μετά από επανειλημμένες εκκλήσεις των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περιμέναμε μια τέτοια αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αναθεώρηση είναι περιορισμένης εμβέλειας και τεχνικής φύσεως, γιατί ε, γενικά υπάρχουν θέματα τα οποία εφαρμόζονται πλήρως. Όμως η πρόταση αυτή θα πρέπει να γεφυρώσει το διακανονιστικό κενό το οποίο υπάρχει σε σχέση με τις ισχύουσες διατάξεις και τις επιλεκτικές τακτικές που ακολουθούν συγκεκριμένες χώρες μέλη σε σχέση με την εφαρμογή του συνόλου του πακέτου. Αυτό μας απασχολεί λοιπόν στον τομέα των αγωγών λοιπά. Όπως υπόθηκε κατά τη διάρκεια και της χθεσινής ακρόασης, έχουμε καθυστερήσει κατά μία αιτία. Είναι λοιπόν καλό να τα κάνει κανείς τα πράγματα σε όσο το ταχύτερο γίνεται, αλλά από την άλλη κάλιο αργά παρά ποτέ όπως λέμε. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση τώρα και θα πρέπει να κλείσει το θέμα αυτό χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, γιατί όπως καταλαβαίνετε και εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι είναι ένα από τα αρκετά σημαντικά θέματα τα οποία έχουμε μπροστά μας. Εγώ έχω στην ουσία βάλει πολύ λίγες συμπληρώσεις στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ελών της Επιτροπής μας, γιατί όπως σας είπα δεν έχουν κατατεθεί πάρα πολλές τροπολογίες. Αυτό θα μας διευκολύνει να παρουσιάσουμε με βάση την δική μου πρόταση τις λεγόμενες συμβιβαστικές. Θα τις προετοιμάσουμε τις συμβιβαστικές νομίζω ήδη από την επόμενη εβδορίση στις συζητήσεις και όπως είπα η οδηγία αυτή είναι περιορισμένου μεγέθους και τεχνικής φύσεως. Οπότε μέσα σε μία εβδομάδα θα επεξεργαστούμε όλες τις τροπολογίες και θα είμαστε έτοιμοι για την ψηφοφορία η οποία θα γίνει την 21η Μαρτίου ε, για την ολοκλήρωση των κανονισμών σχετικά με την εσωτερική αγορά. Αυτό το οποίο είναι ανησυχητικό από δική μου πλευράς τουλάχιστον είναι η θέση την οποία θα ακολουθήσει το Συμβούλιο. Ε, έχουμε ανάγκη την θέση του Συμβουλίου τον Μάρτιο για να ξεκινήσει επιτέλους ο της λίγες τροπολογίας. Περιορισμένης εμβέλειας θα έλεγα, αλλά η θέση του Συμβουλίου είναι πολύ σημαντική και γι' αυτό ε, προσδοκούμε, εν πάση περιπτώσει, να υπάρξει από πλευρά του Συμβουλίου μια τέτοια θέση. Έτοιμη στι 21 Μαρτίου πάντω. όταν προσπαθώ να συντάξω τις συμβιβαστικές τροπολογίες θα λάβουμε υπόψη μας όλες τις προηγούμενες συζητήσεις στην Ήτρε όπως επίσης και τις διαβουλεύσεις τις οποίες κάναμε με τους εμπλεκόμενους τα θαμέλη. Έχει κρίσιμη σημασία για μένα ε, να λάβω υπόψη τη τροπολογία σας και γι' αυτό θα ήθελα αν το επιθυμείτε να μου πείτε ποιες από τις τροπολογίες που έχετε καταθέσει είναι σημαντικές για την ενίσχυση και τη βελτίωση της τελικής μου πρότασης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ως και ο θα ήθελα να τονίσω αυτά που έχω ήδη πει στο παρελθόν. Το έκανα και αυτές. Πιστεύω ότι η αναθεώρηση αυτής της οδηγίας πρέπει να τεθεί σε συνεδρίαση, στις επόμενες συνεδρίε. Ευχαριστώ πολύ. Και ο κύριος Σιλκιώτης. Ε, οι τροπολογίες που έχουν καταδεθεί επιβιώνουν ε, πως υπάρχει μεγάλη ανησυχία και προβληματισμός για τις αρνητικές συνέπειες που θα έχει η προτινόμενη οδηγία για το φυσικό αέριο. Εξού και πολλοί ευρωβουλευτές από διάφορες πολιτικές ομάδες δεν ζητούν απλά αλλαγέ, αλλά τη συνολική απόρριψη της οδηγίας. Η ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς κρίνει πρώτα-πρώτα ως <clears throat> απαράδεκτο το γεγονός ότι οι προτινόμενες αλλαγές στην οδηγία και αναφέρομαι στην Επιτροπή, παρουσιάστηκαν χωρίς καμιά διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και χωρίς εκτίμηση των επιπτώσεων όπω απαιτούν οι κατευθυντήριε γραμμές για την αλλαγή της νομοθεσίας. Αλλά για μας το χειρότερο είναι πως η προτινόμενη οδηγία αποσκοπεί στη χειραγώγηση των κρατών μελών σχετικά με την ανάπτυξη συναγωγών με τρίτες χώρε. Ιδιαίτερα όταν γίνεται προσπάθεια να ελέγξει η Κομισιόν ακόμη και τους αγωγους εξαγωγή εξαγωγής από κράτη-μέλη φυσικού αερού προς τρίτες χώρες. Ε, γι' αυτό λέμε ξεκάθαρα πώ θα στηρίξουμε μια πρόταση η οποία έχει στόχο να ακυρώσει τα κυριαρχικά δικαιώματα και τι εξουσίε των κρατών μελών σχετικά με του όρου εκμετάλλευση των ενεργειακών του σπόρων. Αντί η Κομισιόν να καταθέσει προτάσει, εισηγήσει, να αναλάβει πρωτοβουλίε για να λύσει τα πολλά αδιέξοδα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ενεργειακή τροφοδοσία και ασφάλεια, με την ελόγω οδηγία θα δημιουργήσει περισσότερα νέα προβλήματα τόσο στη λειτουργία των υφιστάμενων αγωγών, όσο και στην άπτυξη νέων αγωγών. Και να φέρω ω παράδειγμα των αγωγών ΙΣΜΕΤ, είναι ο αγωγό που βρίσκεται τώρα σε μελέτη, είναι από την Ανατολική Μεσόγειο, ε, μέσω Ελλάδα και Ιταλία προ την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίο θα μεταφέρει το φυσικό αέριο στο ευρωπαϊκό σύστημα από αυτήν την ε, περιοχή. Είναι για αυτούς τους λόγους που έχουμε ε, τους προβληματισμούς μας. Ε, όμως ε, πριν να κλείσω θα ήθελα κύριε Πρόεδρε και αναφέρομαι σε εσά ω εισηγητή τη εκθέση για το φυσικό αέριο ε, και ω ο πρόεδρο τη Επιτροπή μα, που είναι καθόλου ε, αρμόδια για τα θέματα ενέργεια, να λάβει μια πρωτοβουλία ε, και να ασκήσει πιέσει προ την Τουρκία για να σταματήσει άμεσα τι παράνομε ενέργειε στην Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη, οι οποίε εμποδίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία να ασκήσει τα κυριαρχικά τη δικαιώματα. Το αναφέρω εδώ, διότι συζητούμε για την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου από τη στιγμή που εδώ και μέρες η Τουρκία παράνομα εμποδίζει μια ε, ευρωπαϊκή εταιρεία, την Ιταλική εταιρεία Νένη, να, εισέλθει στην Κυπριακή ΑΟΣ για να πραγματοποιήσει γεώτρηση σε μια περιοχή με τόσο σημαντικά κοιτάσματα φυσικού αερίου, τα οποία μπορούν πραγματικά να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ένωσης. Έχουν γίνει ήδη δηλώσεις από ε, στο ευρωπαϊκό επίπεδο που καταγγέλνουν την παράνομη δράση της Τουρκίας ωστόσο αυτό δεν σταμάτησε την παράνομη και προκλητική τη δράση και ζητούμε ακριβώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει αποφασιστικά μέτρα να σταματήσει η Τουρκία να δερματίσει άμεσα τι πειρατικές και επικίνδυνες ενέργειε. Ε, και γι' αυτό ε, θα ζητούσα και από εσά, κύριε Πρόεδρε, αν μπορείτε να κάνετε μια παρέμβαση για το θέμα, γιατί δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε σήμερα για ενίσχυση τη αγορά του αγρίου και ενδυνάμωση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα όταν έχουμε ακριβώς με, να κάνουμε με τέτοιες παράνομες συνεργίες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Προκειμένου να είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, κάτι άλλο που είναι σημαντικό, θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε με τον εισηγητή και τους εισηγητές οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα θέλουμε να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιπτώσεις εμπειρογνώμονές μας. Και εγώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι. Καλύτερη νομοθεσία, καλύτερη ρύθμιση, η οδηγία. Μπορέσαμε δηλαδή να αντιδράσουμε και να διαχειριστούμε καλή συνθήκες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης από τρίτες χώρες. Κύριε Κόπελ. προτείνεται συνθήκες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης από τρίτες χώρες. Κύριε Κόπελ. Προτείνεται να μην υπάρχουν εξαιρέσεις. Αυτές όμως τις εξαιρέσεις τις χρειαζόμαστε, γιατί για να μπορέσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι πρέπει ε, απομονωθούν από τις διαδρομές της Γκάσπρομ. από την Γκάσπρομ. Και όχι μόνο τους Ισπανούς και τους Ιταλούς και κάποιους Γάλλους και κάποιους Γερμανούς. όλοι αυτοί πιαστικά είναι καθαρά ελεγχόμενοι από τους δυνατότερους. Βλέπουμε σήμερα τους ε, Βουλγάρους οι οποίοι διαμαρτύρονται και έχουν δίκιο για την κατάσταση. Και πραγματικά εμείς σαν ε, Ευρωπαίοι ε, εκπρόσωποι των χωρών της Δυτικής Ευρώπης θα πρέπει λίγο να συνειδητοποιήσουμε τι συμβαίνει. Ευχαριστώ που μου ξαναδίνετε το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Τούρμες, είναι απαράδεκτο. Μία από τις μεγαλύτερες ε, αυστριακές ε, επιχειρήσεις ε, τις ε, παρουσιάζετε με έναν τόσο δυσμενή τρόπο. Προσπαθείτε να ποινικοποιήσετε δραστηριότητες που δεν έχουν τίποτα το παράνομο. Πρόκειται για μια επιχείρηση η οποία είναι στο χρηματιστήριο της Αυστρίας και φυσικά και υπάρχουν διαδρομές από την Ρωσία και φυσικά και γνωρίζουμε ε, την επιχείρηση Gazprom και το ρόλο της, αλλά πραγματικά πρέπει, επαναλαμβάνω, να βρεθεί πολιτική λύση έτσι ώστε η Ρωσία να μπορέσει να έχει μια διαφορετική δράση. Αυτό που όλοι χρειαζόμαστε και νομίζω συμφωνούμε όλοι, είναι να υπάρχει ασφάλεια για τον Ευρωπαίο καταναλωτή, να υπάρχει εφοδιασμός με ασφάλεια. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις πραγματικές ανάγκες της Ευρώπης, των πολιτών της Ευρώπης, όταν μιλάμε για ενεργειακή ένωση. Αυτή θα πρέπει να είναι η στόχη μας. Πρόεδρος. Να να είμαστε ήσυχοι όταν μιλάμε για το θέμα αυτό. κύριος ε, Ρούμπιχ. Ίσως είναι και όποια απόψεις. σε συμβάσεις, τα υπάρχοντα έργα και πραγματικά το πραγματικό διακύβευμα είναι μάλλον στην Νότια Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι μιλάμε για βαλτικές χώρες και ξέρουμε τις πάρα πολύ μεγάλες αντιρρήσεις στο μεγάλο έργο, αλλά πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί είστε τόσο επικριτικοί. Έχουμε και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εχθές ξεκίνησε ο τριμεριουμέ με, με το πακέτο για την καθαρή ενέργεια. Και κάθε φορά που οι θέματα που αφορούν την ενέργεια. Είστε πάρα πολύ χρήσιμοι. Δεν συμφωνούμε πάντα μαζί σας. Ευθυντά. Thank you very much, uh, Mr. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δώσατε την δυνατότητα να σχολιάσω τις τροπολογίες. Καταρχάς να υπενθυμίσω. Υπάρχει λόγος τώρα να επαναλάβω αυτά τα οποία σας είχα πει στην τελευταία μας συνάντηση. Θα ήθελα να συγκεντρώσω την προσοχή μου σε μεμονωμένες τροπολογίες. Σήμερα το πρωί εξέφρασε την άποψη ότι δεν έχει υπάρξει μελέτη επιπτώσεων για την συγκεκριμένη πρόταση. Εδώ να μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω ότι που δεν έχει περάσει από μελέτη επιπτώσεων παραβιάζουμε τους κανόνες αυτούς. Με την πρόταση αυτή βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη θα έλεγα κατάσταση. Ασία να μπορέσουμε να εξετάσουμε όλες τις μεμονωμένες τροπολογίες, τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να, όταν συζητήσουμε την τελική πρόταση που θα καταθέσουμε στην Επιτροπή. Τις ακούστηκαν να υπογραμμίσω λοιπόν κάποια σύντομα τελικά σημεία. Για την τρίμηνη μεταφορά. Είναι κάτι το προφανές θα έλεγα το θέμα αυτό για το σύνολο της μεταφορά ε, της ισχύω της ρύθμισης αυτής είναι προφανής και απαραίτητη και για τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες. Αν μιλάμε σαν παράδειγμα για το εμπόριο κινέζικων παιχνιδιών, ιαπωνικών αυτοκινήτων ή αμερικανικών υπολογιστών, είναι προ... και αυτό είναι ένα επιπλέον ε, πρόβλημα. Όμως στο συγκεκριμένο κανονισμό δεν θα πρέπει να ονοματίσουμε. Εμείς κάνουμε διάκριση ανάμεσα στα υπάρχοντα προγράμματα και στα υποπροετοιμασία τα μελλοντικά είναι σαφές ότι ε, έχουμε ανάγκη για το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα τέτοιο κανονισμό. Και γι' αυτό τη διευκρίνηση αυτή μετά από συζήτηση με τους Σκιώδης και θα προσπαθήσουμε να λύσουμε κάποια συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν. Και χθε είχαμε την δυνατότητα να τα συζητήσουμε αυτά με ε, υψηλούς εκπροσώπους από την Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας προτείνω την επόμενη εβδομάδα να υπάρξει μια συνάντηση, μάλλον να στείλουμε τις προτάσεις προς τους σκιώδεις ε, κάποιες συμβιβαστικές τροπολογίες τις ομιλίες σας, ενισχύει και βελτιώνει τις ιδέες που περιλαμβάνονται στην αρχική μου πρόταση. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τις συζητήσεις με αυτή την βάση. Και να μην ξεχνάμε ότι θα ψηφίσουμε την ερεσμία από πλευράς μας. Περιμένουμε λοιπόν και από τη Βουλγαρική Προεδρία να παρουσιάσει την κοινή θέση του Συμβουλίου και να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τον τριμερή διάλογο στις αρχές Απριλίου. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας, συνάδελφοι, και περνάμε τώρα στο... Και αυτό είναι αντικείμενο προφορικής ερώτησης. Βρίσκεται υπό προετοιμασία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε το θέμα των τεχνολογιών DLT και των συστημάτων blockchains. Αυτό το θέμα απασχολεί το τύπο και διάφορους παραγόντες. Το, το πολύ περίπλοκο σύστημα που υπόσχεται πολλά όμως και ε, πιστεύω ότι η προσέγγιση μας θα επιφέρει διευκρινήσεις. Οι τεχνολογικές ε, εξελίξεις θα συζητηθούν ε, στα εργαστήριά μας. Θα προσπαθήσω να βρω το εξοπλισμό. Έχουμε το θέμα των cloud και της αποκέντρωσης του εξοπλισμού και τώρα δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να χρησιμοποιήσουν και αποκεντρωμένο εξοπλισμό και αποκεντρωμένα δεδομένα. Αυτό ε, υπόσχεται πολλά ως προς οι τεχνολογίες DLT. Πρόκειται για διάφορες ε, τεχνολογίες με κοινά χαρακτηριστικά. Ο στόχος αυτού του ψηφίσματος ε, είναι να δείξει ότι οι εφαρμογές των DLT και των blockchain δεν είναι μόνο το bitcoin, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, ο ενεργειακός τομέας μπορούν ε, να εφαρμοστούν πολύ της φορολογικής διαφυγής. Οι τεχνολογίες αυτές πρόκειται ουσιαστικά για κατανεμημένες βάσεις δεδομένων με κρυπτογραφικές υπογραφές. Υπάρχει και μια πολύ σημαντική συμβάλλουν αυτές οι τεχνολογίες και τη χρηματοδότηση των και των ατόμων τεχνολογίων. Χρειάζονται φυσικά διευκρινήσεις ε, και σε νομικό να συμβάλλουν στην διαλειτουργικότητα, στην τυποποίηση ε, των ε, κανόνων σε αυτούς τους τομείς. Είναι σημαντική φυσικά τα συστήματα blockchains. Πρέπει να υπόκεινται σε ρυθμίσεις της χρήσης τους επιπλέον θα ήθελα να τονίσω την εξαιρετική συνεργασία που η ομάδα μου είχε με τις ε, Γενικές Διεμφύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεργαστήκαμε και με ε, πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Ευχαριστήσουμε να είμαστε ευγνώμονες για αυτές τις πολύ σημαντικές συνεργασίες που θα συμβάλλει στην εξέλιξη της ψηφιακής οικονομίας. Νομίζω ότι η Ευρώπη μπορεί να είναι ηγέτη σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια. Ευχαριστώ την εισηγήτρια, την κυρία Καηλή, για την οργάνωση των workshop το τελευταίο έγινε σήμερα το πρωί, αλλά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον που πραγματικά ακούσαμε εμπειρογνώμονες οι οποίοι μας εξήγησαν και μας βοήθησαν. Πρόκειται για μια επανάσταση. Άλλοι λένε ότι είναι εξίσου σημαντική με την ε, δημιουργία του διαδικτύου. Άλλοι λένε ότι θα αλλάξει πολλά, αλλά όχι τόσο πολύ σημαντική επανάσταση. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε αυτή την εξέλιξη, να στηρίζουμε τις νέες τεχνολογίες. Εγώ συμφωνώ με την πολύ σωροπημένη προσέγγιση της εισηγήτριας. Θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η Ευρώπη μία ήπειρος που θα είναι πολύ για την Επιτροπή μας. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργούμε αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο να λειτουργεί στην Ευρώπη. Αν έχουν προετοιμαστεί σωστά για αυτές τις νέες τεχνολογικές λύσεις. Παραδείγματο χάρη των ηλεκτρονικών υπογραφών αναγνωρίζονται. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν τα κράτη-μέλη να συνειδητοποιήσουν ότι δεν πρόκειται μόνο για τα κρυπτονομίσματα, γνωστά ιδιαίτερα μέσω του bitcoin ή εδώ και λίγο καιρό για να εξετάσουν όλες τις πρακτικές εφαρμογές της τεχνολογίας blockchain. Και από ό,τι φαίνεται σε σταθμούς ανεφοδιασμού για τις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων κτλ. Ας κάνουμε με το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής και στηρίζουμε τις περισσότερες προτάσεις. Πρόκειται για ένα δύσκολο και περίπλοκο θέμα και βέβαια οι τομείς ε, που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν αυτές οι τεχνολογίες. Θα προσέθετα στους δύο τομείς που αυτών που δεν συνάδουν με το EGTR. Θα ήθελα να ζητηθεί νομική ότι είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες της Ευρώπης να μπορούν να μετακινηθούν και να βάλουν το ψηφοδέλτιο στην κάλπη.